Καλησπέρα. Καλημέρα, συγγνώμη, <laughs> κυρίες και κύριοι. Καλώ ήρθατε στη συνεθρίασή μας. Έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε διάφορες ψηφοφορίε. Οπότε σας ευχαριστώ που ήρθατε στην ώρα σας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Πριν όμως ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία, πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ο κύριος Ομερζέ δεν θα μπορέσει να έρθει και ε, πρόκειται για το σημείο 16 στην ημερήσια διάταξη, έτσι, οπότε αναβάλλεται για μια άλλη συνεδρίαση. Εντάξει, ωραία. Το ξέρετε. Και οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ενημερώνονται ότι δεν θα εξετάσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η γνωμοδότησή του θα συμπεριληφθεί σε μία από τις συνεδριάσεις μας του Δεκεμβρίου. Άρα δεν θα έχουμε το σημείο 16 σήμερα στην ημερήσια διάταξη και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Η πρώτη μας ψηφοφορία είναι ο μηχανισμός για την άρση νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Είναι νομοθετικός φάκελος αυτός για τον οποίο είμαστε εμείς αρμόδιοι επί της ουσίας. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος ματές Φαν Μίλτεμπερκ, ο οποίος παρουσίασε στις 15 Οκτωβρίου το σχέδιο εκθεσής του. Έχουμε 119 τροπολογίες που υποβλήθηκαν και 11 συμβιβαστικές μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η Ένβη γνωμοδοτεί και έχουν και εκείνοι τις δικές τους προτάσεις. Πριν περάσουμε όμως στην ψηφοφορία θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και κάποιες πολιτικές ομάδες μου είπαν ότι οι σκιώδεις θα έχουν κάτι να πούνε. Λοιπόν, κύριε Φαν Μίλτεμπεργκ, παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδες εισηγητές για την επικοδομητική τους προσέγγιση και ελπίζω ότι και το ΕΛΚ τελικά θα υπερψηφίσει αυτή την έκθεση, ξέροντας ότι έχουμε συζητήσει πολύ για την εθελοντική βάση αυτού του μηχανισμού. Θα δούμε. Θέλω να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, η νομική υπηρεσία, γραμματεία, PRS, όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θέλω να τους ευχαριστήσω ειλικρινά και ελπίζω ο κύριο Σάλβα να είναι τόσο επικοδομητικό όπω ήταν και στην πρώτη συνάντηση του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Ζέλε τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φαν και τους λοιπούς συνεισηγητές. Ήταν πολύ ζωντανή η ανταλλαγή απόψεων για τον κανονισμό αυτόν. Ένα σημείο και το ανέφερε ο κύριος ε, συνάδελφος, δεν σε ένα σημείο δεν εξασφαλίστηκε συμφωνία. Όπως ξέρετε εξ αρχής, η δική μου θέση ήταν ότι έπρεπε να υποστηριχθεί η περσινοριακή συνεργασία. Άλλωστε αυτό σημαίνει συνοχή για μένα, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους παρά τα εφιστάμενα ε, εθνικά σύνορα μεταξύ τους ε, περιφέρειες διαφορετικών κρατών. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα σύνορα, είναι τα διαφορετικά νομικά συστήματα. Και αυτό σημαίνει ε, πολλές φορές ότι δυσκολεύει ιδιαίτερα η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Και έτσι, γι' αυτό θεωρώντας ότι είναι απαραίτητη η διασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία και με την ύπαρξη των, του δικτύου των, της διασυνοριακής συνεργασίας που ήδη υπάρχει, πλέον τέτοιου είδους ε, ενώσεις ε, που μπορούμε και πρέπει να υποστηρίξουμε γιατί επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται ε, εντατικά για να υποστηρίξουν το έργο αυτό. Ένα παράδειγμα θα ήταν η έγκριση ενός μιας γραμμής λεωφορείου όπως ε, αυτό, αυτή η γραμμή που θα συνέδεε τη Φραγκφούρτη στον Όντερ και το Ζήριου ε, στην ε, Πολωνία που πέρασαν πέντε χρόνια για να εγκριθεί. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα ακόμα και η ίδρυση μιας ε, γραμμής λεωφορείου μεταξύ δύο πόλεων που είναι πάρα πολύ κοντά αλλά τις χωρίζουν εθνικά σύνορα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε όπως είπαμε διαφορετικά εθνικά ένομα συστήματα, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα για τις περιφέρειες να επιλέγουν μόνες τους με ποιο τρόπο θέλουν να εξασφαλίσουν τη συνεργασία αυτή. Έχουμε και από τις εθνικές βουλές και από τις τοπικές ε, πρωτεύουσες ε, επιστολές λάβει ε, που εκφράσουν ανησυχίες σε σχέση με την εθνική κυριαρχία. Υπάρχουν φόβοι δηλαδή ότι απειλείται η εθνική κυριαρχία. Αυτό όμως δεν ισχύει παραμένουν κυρίαρχα τα κράτη, τα κράτη αποφασίζουν. Αλλά πρέπει να επιτρέψουμε, να υποστηρίξουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν, εάν περιέλθει σε όρους ε, ε, εφαρμογής εκούσιας από τα κράτη-μέλη, πολύ φοβούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και τον κίνδυνο των παρεξηγήσεων και παρερμηνιών, αλλά και τη στενοκεφαλιάς που μερικές φορές εμποδίζει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Και γι' αυτό θα ήθελα να είναι πιο δεσμευτικό το νομοθέτημα αυτό. Όπως είπα, δεν παρεμποδίζεται καθόλου η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, δεν περιστέλλεται καθόλου η εθνική κυριαρχία των κρατών, απλώς επιτρέπεται στις περιφέρειες πέραν των συνόρων να συνεργάζονται εκεί που θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να συνεργάζονται. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε συμβαστική λύση εφόσον δεν ε, περιοριζόμαστε σε όρους ε, εκούσιας εφαρμογής. Ευχαριστούμε κύριε Ζελέ. Κατ' εξαίρεση, ε. γιατί δεν θα ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση, όχι σήμερα. Είμαστε στην ψηφοφορία. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στον κατάλογο ψηφοφορίας παρακαλώ. Και επιτρέψτε μου σήμερα να είμαι λίγο πιο αργή γιατί έχουμε δύσκολες υποθέσεις. Δεν θα βιαστώ, χρόνο έχουμε, οπότε ας πάρουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε για την ψηφοφορία. Για το ΕΛΚ. Έχετε 13 μέλη παρόντα εδώ. Ξέρω, είσαστε πολύ δραστήριοι, αλλά να ξέρετε ότι μόνο 12 μπορούν να ψηφίσουν, έτσι, να συμμετέχουν στην πληροφορία. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση, δεν την ακούσαμε. Ο κύριος Όλμπριχτ θα είναι παρατηρητής. Ωραία, καλώς. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία με τη συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε, να δούμε πώς έχει κατάσταση στην αίθουσα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. 18 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίθηκε λοιπόν η συμβαστική 5 και πάμε στην τροπολογία 62. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε για την 67. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 9 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε μαζί μπλοκ διάφορες τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ, ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκαν. Τώρα, Τροπολογία 82. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τότε, να ελέγξουμε. Μπορεί να έκανα λάθος. Ναι, 82. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Ναι, απορρίφθηκε. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95 και 96 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα μαζί, block vote. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103. Συγγνώμη, μαζί ήταν. 102 και 103 ήταν μαζί. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία παρακαλώ. 102 και 103. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε μαζί τέσσερις τροπολογίες, 24, 25, 26 και 27. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δύο τροπολογίες μαζί, 114 και 115 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβιβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην NV1 στις ιδεολογικές σκέψεις υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Να ελέγξουμε, ναι, να ελέγξουμε για την NV1 στην αιτιολογική σκέψη 2α. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. NV2 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω όλα θα ελέγξουμε καλύτερα. Για τη συμβαστική τροπολογία 2, ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 51. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος απορρίφθηκε. Με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 52. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε. Συμβαστική τροπολογία 4, λοιπόν, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τώρα, τροπολογία αριθμός 61. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Αλέξουμε 61. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Λοιπόν, εγκρίθηκε η έκθεση. Και τώρα πρέπει Παρακαλώ. Αποχή. Για μένα αποχή, βεβαίως. Καλώς. 14 υπέρ, ένα κατά και 15 αποχές. Έχει γίνει πλέον δεκτή. Α. Ζητώ συγγνώμη, μπερδεύτηκα λέει η πρόεδρος. Νόμιζα ότι δεν έγινε δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε για τη διαπραγματευτική εντολή. Ποιοι είναι υπέρ του να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας μέχρι τώρα. Ψηφίζουμε τώρα την επόμενη γνωμοδότησή μας για το πρόγραμμα InvestEU. Η συγγήτρια κυρία Βέσφαλ παρουσίασε τη γνωμοδότησή της το Σεπτέμβριο. 245 οι τροπολογίες. Συ 21 συμβιβαστικές υπεύθυνε επιτροπές από κοινού, η ΕΚΟΝ και η μπάτζετ. Θέλετε το λόγο κύριε Βέσφαλ. Ναι, όντως και πολύ σύντομα πριν περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Είχα επισημανεί και στην παρουσίαση της έκθεσης ότι με ενδιαφέρει να διαγράψουμε αυτό το Member State Compartment, διότι η συζήτηση έγινε βεβαίως μέσα στην μικρή αυτή γνωμάτευση ε, με βάση το πώς εμείς τοποθετούμαστε, το πώς αντιμετωπίζουμε τη θέση μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που με στήριξαν. Πρέπει να βγει αυτό το Member State Compartment, επαναλαμβάνω, και περιμένω να δω τι αποτέλεσμα θα προκύψει. Για μένα ήταν μια κόκκινη γραμμή, γιατί πρόκειται για μια αλλαγή συστήματος. Η διαρθρωτική πολιτική είναι διαρθρωτική, πολιτική είναι πολιτική των ενισχύσεων, της υποστήριξη, έτσι πρέπει να μείνει και όπως έχω ξαναπεί δεν πρέπει στον βωμό του έτσι να θυσιαστεί η περιφερειακή μας πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες λοιπόν. Ανάλογα με την ψηφοφορία θα δούμε πώς θα πάμε με τα υπόλοιπα θέματα. Θα ξεκινήσουμε με την 12 και την 127 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί τώρα ξεκινάμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος 12 και 127 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Οπότε περνάμε τώρα στην 109. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Έντεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές το ίδιο δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 163. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 16. Απερίφθη. Δεκαεπτά υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 18 υπέρ. Μαζί με την 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τέσσερα και εβδομήντα ένα υπέρ κατά αποχές απερίφθη δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 107 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 110 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή πηγαίνουμε στην 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 111. Έχει καταπέσει. Γιατί απερίφθηκε 124. Το ίδιο και για την 112. Και πηγαίνουμε στην 148. Ταυτόσιμες. Νομίζω ότι το 112 δεν είναι το ίδιο με το 111, λέει η κυρία Κρέλ. δεν είναι ταυτόσιμες εντελώς. Κανονικά τις ψηφίζουμε ξεχωριστά. Αλλά και οι δύο έχουν καταπέσει, γιατί απορρίψαμε τις προηγούμενες. Συγγνώμη λέει η κυρία Κρέλ. 148 τώρα και 149 ταυτόσιμες ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. Δεκ, δεκτές.

Οπότε θα ψηφίσουμε τώρα την τελευταία προσθήκη mainstreaming του κλίματος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 47 λέει η πρόεδρος. υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. οκτώ καταπίπτει. Εκατόν τριάντα δύο. Συμβιβαστική τρία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 154. Υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 154. Τέλος. Απερίφθη. Εκατόν Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 155 υπέρ. Εξ, κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15, 159 και 160 ταυτόσημες ψηφίζονται από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 162 υπέρ. Κατά Αποχές. Δεκτή. 166. Καταπίπτει. Καταπίπτει και η 165. 169 καταπίπτει. Πάμε λοιπόν στο 174. Καταπίπτει και αυτή. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 180. Τέλος. Απερίφθη. 181. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 184. Υπέρ. Κατά αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 190. Υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 190. Υπέρ Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ναι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Μεγάλη έκπληξη για μένα. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να σηκώνετε πάντα τα χέρια σας. Όχι, το ένα, το ένα παρακαλώ. Αλλά να τα σηκώνετε εγκαίρως. Γιατί κάνω λάθη και λείπουμε πολύ. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 194 υπέρ κατά αποχές, α, ε, αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 196 έχει καταπέσει. 197 έχει καταπέσει. 217 έχει καταπέσει. Η 81 έχει καταπέσει. 131 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. η 479 καταπίπτει 215 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε τη 215 ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται. 80 καταπίπτει. 199 και 200 τώρα, ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές απεριφθεί. 82 και 83 πάλι ταυτόσιμες. Α, όχι, καταπίπτουν. Καταπίπτουν. Και περνάμε. Στη 201. 1 Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 202 καταπίπτει. Έτσι δεν είναι. Και 203 καταπίπτει. Διακόσια την ψηφίζουμε. Και τη 202. Όχι. 203. Όχι, είναι πολύ παράξενος ο καταλογός μου. Παρακαλώ, 203 υπέρ. 203 κατά απόχες και απεριφθεί. 204 υπέρ κατά απόχες απεριφθεί. 205 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 206 καταπίπτει όχι την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απερίφθη 207-208 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 209 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 210 211 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2.13 υπέρ κατά αποχές και νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Ελέγχουμε την 2.14. Όχι, λυπούμε. 2.13. 2.13 ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Σαφώς. Δύο δεκαέξι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο δεκαοχτώ υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Δύο δεκαεννέα υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 2.20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2.23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ταυτόσιμες 26, 2.24, 2.25 20 και 2.25 τρεις είναι 26, 2.24, 2.25 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε 2.25 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Δεκαπέντε υπέρ. Πώς γίνεται αυτό. Και απερίφθη, ναι. Ένας δεν ψήφισε. Απερίφθη. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27-2, 229 ταυτόσημε υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. 2.30 καταπέπτει, 2.31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 232 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 232 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 237 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 238 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 239 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 240 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 241 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 242 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 243 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 244 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ, α, καταπίπτει. 77 επίσης, 78 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Καταπίπτει. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Α, καταπίπτει γιατί 12. 97 ναι. τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 97. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Πρέπει να με απολύσετε σήμερα, λέει η πρόεδρος. Πάω πολύ γρήγορα, μήπως. Συμβαστική 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, που είναι ίδια με την 103 και την 104. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 105, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Θέλετε το λόγο, κύριε Βέσφαλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας. Πραγματικά δεν ε, το θεωρούσα σίγουρο, αλλά δεδομένου ότι κερδίσαμε σε αυτή την πρώτη ψηφοφορία, σας ευχαριστώ πολύ. Γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής, οπότε σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας στην ψηφοφορία. Τώρα, συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο μας θέμα, την επόμενη ψηφοφορία για σήμερα, που είναι γνωμοδότηση για την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Η συγκητής είναι ο κύριος Φαν Μίλτεμπεργκ, ο οποίος μας παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησής του τον Οκτώβριο νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. 128 τροπολογίες είχαμε. Και υπάρχουν και διάφορες συμβαστικές. Έτσι θέλετε μήπως το λόγο, κύριε Φαν Μίλτεμπεργκ. Ναι, ευχαριστώ. Δυστυχώ είναι ένα επίμαχο ζήτημα, οπότε πράγματι είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συμβαστικές προτάσεις. Προσπάθησα, έχουμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές τροπολογίες που παραμένουν και παραμένουν προς, και πηγαίνουν προς κάθε κατεύθυνση. Οπότε ευχαριστώ και πάλι τη στήριξη που είχα από τους Σκιώδες και την ε, Γραμματεία. Κάποιες σεβαστικές προτάσεις έχουμε και ελπίζω να καταλήξουμε, να έχουμε και γνωμοδότηση στο τέλος για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε ως Επιτροπή με την γνωμοδότησή μας ε, τις αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές που είναι η προπολογισμού και συνταγματική. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να έχουμε γνωμοδότηση σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Οπότε αρχίζουμε την ψηφοφορία και ξεκινάμε με την τροπολογία αριθμός 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 40 και 41 που είναι ίδιες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 42. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 43. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος, απορρίφθηκε. Σαράντα τέσσερα τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σαράντα πέντε. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 49 τώρα. 50, 52, 53, 54 και 55. Μαζί τις ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Όλες. Τροπολογία 48 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. 56 λοιπόν υπέρ. Α, θέλετε να το λόγο. Παρακαλώ κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ. Προτείνει ο Σκιώδης εισηγητής μια προφορική τροπολογία στη μέση του κειμένου που σημαίνει ότι το κείμενο θα λέει ελευθερία γνώμης και έκφρασης περιλαμβάνοντας και την ελευθερία τύπου ε, συνεταιρίζεστε Αυτά λέει το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία στην τροπολογία μας 56, σωστά? Σωστά. Είναι κανείς κατά της προφορικής αυτής αλλαγής? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν με την αλλαγή αυτή, την 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 57. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 58. Δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια καλά. Λοιπόν, μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. Πρέπει να βλέπω τα χέρια σας, να σηκώνετε καλά τα χέρια για να τα βλέπω.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 Τροπολογία 68. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71. Υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε 71 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος, εγκρίθηκε. Εβδομήντα δύο τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 και 77 που είναι ίδιες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78, 79 και 80 που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για αυτές τις τρεις, 78, 79 και 80. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογίες 81 και 82 που είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 83-84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. με την προφορική τροποποίηση. Α, ναι, παρακαλώ κύριε Φαρμίλτεμπεργκ. Στο κείμενο της συμβαστικής αυτής, οι σοσιαλιστές το ζήτησαν και προτείνουμε να διαγραφεί η τελευταία πρόταση που αρχίζει από εκεί που λέει ότι η Επιτροπή μπορεί επίσης να λάβει υπόψη της τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται ε, στην προσχώρηση. Αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Είναι σαφές για όλους. Έχετε πάρει την προφορική αυτή τροποποίηση, την έχετε, το ακριβές κείμενο. Καλώς τότε. Συνεπώς, είναι κανείς κατά της τροποποίησης της προφορικής. Ωραία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 5 με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 102 και 103. Που... Αυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθησαν. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Και είναι μαζί 106-107. Χωριστά η 106 υπέρ κατά. Αποχές απεριφθεί. 107 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά. Αποχές και απεριφθεί. 108 υπέρ κατά Αποχές και εγκρίνεται. 112. Όχι. Ναι. Περκατά. Αποχές και εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές απερίφθη 115 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται 117 υπέρ όχι καταπίπτει Ε, με συγχωρείτε, λέει η κυρία Μιχαήλova. 115, 117, 118, 116 καταπίπτουν. Όλες αυτές έχουν καταπέσει. Και πάμε στην 3 και την 119 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Α, και την 120 επίσης. Τρεις, τρεις οι τροπολογίες. 119, 120 και νούμερο 3 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν. Να επαληθεύσουμε. Την 3, ε, την 119, την 120 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 121. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές 123 υπέρ κατά Αποχέ και απερίφθη. 124 κατά αποχές και απερίφθη. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά άποχες και εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη. 127 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 128 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές και περίφθη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη. 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 29 ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 καταπίπτει. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές τριάντα επτά υπέρ κατά αποχές απερίφθη 38 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται και Τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Μπορώ να διατυπώσω μια ερώτηση, παρακαλώ βλέπω ότι ο εισηγητής ο ίδιος καταψήφισε την έκθεση. Διατηρεί την ε, υπογραφή του ή, ή αναλαμβάνει τις συνέπειες. Απάντηση. Κοιτάξτε, πολιτικά για μένα είναι απαράδεικτο. Γιατί ε, ψηφίσαμε να παίρνουμε, διαδικασ... παίρνουμε αποφάσεις μόνο με την ομοφωνία, δηλαδή με διαδικασία ισοδύναμη με αυτή του άρθρου 7. Αποσύρω λοιπόν το όνομά μου από αυτή την έκθεση γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ να καταθέσω γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού με αυτές τις διατάξεις. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση και για την απάντηση. Άρα αποσύρουμε το όνομά σας από την γνωμοδότηση καθώς είναι εγκριθήσα ωστόσο, θα κατατεθεί στην ε, αρμόδια καθήλυνη επιτροπή με το δικό μου όνομα από τη θέση της Προέδρου εκ μέρους της Επιτροπής μας. Στην επόμενη ψηφοφορία. Ενδιαφέρουσα φαντάζομαι πως και η πρώτη. Αλλά είναι η τελευταία για το πρωινό μας σχέδιο γνωμοδότησης, πρόγραμμα διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. προϋπολογισμών και οικονομική είναι οι καθήλυνα αρμόδιες. Έχουμε 152 τροπολογίες με μεγάλες αποκλήσεις οι αρχικές θέσεις στο κείμενο της γνωμοδότησης. Λιγότερες οι συμβαστικές. Αναγκαστικά θα ψηφίσουμε όλες ή τις περισσότερες από τις τροπολογίες μας εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η συγκήτρια. Ευχαριστώ λοιπόν τους Κιώδης ε, και περνώ στην ψηφοφορία χωρίς καθυστέρηση. Τροπολογία 71 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συναφής τώρα τροπολογίες. 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70, συναφείς μεταξύ τους, on block, υπέρ, κατά, αποχές και απερίφθησαν όλες. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. 12 υπέρ. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 90 ηλεκτρονικά, άρχεται. Πέρας, απερίφθη. Ογδόντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 94 υπέρ. Κατά. Απεριφθεί. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 είναι ταυτόσιμη. Εντάξει, λυπάμαι, το ξέχασα. Και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108, ε, 105 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 106 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 107 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 108 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 109 υπέρ προφορική Υπάρχει κανείς κατά της προφορικής. Όχι. Με την προφορική λοιπόν, την 109, υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε 109. Ελέγχουμε. Και πέρας. Δεκτή. 110. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εκατόν δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 111 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 114 116, 117 και 122 συνδεόμενες τροπολογίες από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 115. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συνδεόμενες τροπολογίες τώρα 123, 124 και 125. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεκτές μάλλον. Συνεχίζουμε τώρα με την 126. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθεια. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθεια. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθηκε αυτή. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε όλο και λιγότεροι. τριάντα 135 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 140 έχει αποσύρθει. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 και 41 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές δε, απερίφθη. 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 53 υπέρ κατά αποχές αδεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61 Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονικός έλεγχος για την 7. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. τέσσερα. υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική δέκα. υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εννέα. υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απερίφη 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. Η γνωμοδότηση σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας και έτσι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Πήγαμε πιο αργά από ό,τι συνήθως, αλλά ήταν σημαντικό να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Να συνεχίσουμε παρακαλώ, γιατί έχουμε αρκετά θέματα ακόμα στην ημερήσια διάταξη. Προτείνω το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη να είναι ή μάλλον το επόμενο θέμα στη μέση διάταξη που είναι η αποστολή αντιπροσωπείας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ίσο Ρεουνιόν στη Γαλλία που έλαβε χώρο το επομενο θεμα στη μεση διαταξη που ειναι η αποστολη αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη στην ισο ρεουνιον στη γαλλια που ελαβε χωρο το σεπτεμβριο να αναβληθεί γιατί έχουμε ήδη την γραπτή έκθεση για την αποστολή αυτή αλλά ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποιες κάπως δυσάρεστες καταστάσεις στην περιοχή και καλό θα ήταν να έχουμε εδώ και τον κύριο Μερζέ μαζί μας για να μας ενημερώσει για την τρέχουσα κατάσταση. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν θα αναβληθεί η συζήτηση για αυτό το θέμα και θα το συζητήσουμε όταν θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μερζέ. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε. 1η Ιουνίου 2018 παρουσίασε το πακέτο μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή γεωργική πολιτική που περιλαμβάνει πρόταση για θέσπιση κανόνων σχετικά με τη στήριξη στρατηγικών σχεδίων που θα καταρτιστούν από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, τα στρατηγικά σχέδια για την κοινή γεωργική πολιτική προβλέπουν διατάξεις για διαφόρων ειδών παρεμβάσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από τις χώρες μέλη μέσω των άμεσων ενισχύσεων, ε, μέτρων ενίσχυσης της υπαίθρου και τομεακά σχέδια. Έχουμε ορίσει τον κύριο Ροπέ ως εισηγητή μας για την γνωμοδότηση, συντάκτη συντάκτης γνωμοδότησης και σήμερα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο κύριο Ροπέ και μετά στους σκιώδες εισηγητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Όπως είπε και η Πρόεδρος, σας παρουσιάζουμε τη γνωμοδότηση της ε, δικιάς μας Περιφερειακής Επιτροπής. για αυτό το σχέδιο. Και ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου, γιατί μαζί τους αξιολογήσαμε την κατάσταση, εκτιμήσαμε πώς έχουν τα πράγματα στον γεωργικό τομέα και ποιες είναι οι εξελίξεις και στην Υπαθρό και καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις, 87 ουσιαστικά, δεν και λίγες. Πρόκειται για διαφορετικές συστάσεις και προτάσεις να βελτιώσουμε τον, τους κανόνες αυτούς. Θα είχατε την ευκαιρία να τα δείτε όλα αυτά, οπότε ελπίζω να μου δώσετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και όταν τα ακούσω όλα αυτά τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και παρετέρω και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε, γιατί η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη. Να δούμε δηλαδή με τι θέση θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, ώστε να προτείνουμε και στην Επιτροπή Γεωργίας και ανάπτυξη της Υπέθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Είναι ένα σημαντικός τομέας, όχι μόνο για τη Γεωργία, αλλά και για την ε, ζωή στην Ήπεθρο και στις περιφέρειες. Πολλές πτυχές έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των περιφερειών, με τη βιωσιμότητά τους. Και είναι πραγματικά κρίμα που η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως αρνητική. Το πρόγραμμα το οποίο περικόπτεται περισσότερο οικονομικά είναι ακριβώς αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο ύπεθρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει τη δημοτικότητά της και γι' αυτό έχουν περικοπεί τόσο πολύ τα κονδύλια. Κατά το 1 τέταρτο περίπου. Και αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις η Ευρώπη, το Brexit και άλλες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την επιστημονική έρευνα Οπότε γιατί είναι η ύπεθρος αυτή που πρέπει να επομιστεί το βάρος αυτών των νέων προκλήσεων. Όταν βλέπουμε και ποιο είναι το επίπεδο εσόδων στην ύπεθρο, διαπιστώνουμε ότι είναι το ίμιση των αντίστοιχων στις αστικές περιοχές. Γιατί λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα έσοδα των περιφερειών της Υπέθρου. Χαίρομαι πάντως που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαφορετική στάση από αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε ελπίζω να καταφέρουμε να επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα και να επιμείνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περικοπές στα γεωργικά κονδύλια για την ε, νέα περίοδο. Επίσης είδα κάπως δυσάρεστο που είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση της συγχρηματοδότησης. Οι φορείς που έχουν ε, δραστηριότητες, συνεπώς θα πρέπει να βρουν το διπλάσιο ποσό για να μπορέσουν τώρα να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματά τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες που δίνονται εδώ. Στις πλούσιες χώρες μπορεί να εφαρμόζονται επιτυχώς αυτά τα προγράμματα, αλλά στις λιγότερο αναπτυγμένες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση και δεν υπάρχουν ε, ίδια ήδη πόροι, ε, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Οπότε αυτό που θα γίνει είναι ότι δεν θα υπάρχουν πόροι στις στοχές χώρες και θα ανακαταναμεθούν στις πλούσιες τα ποσά αυτά. Εγώ λέω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις σημερινές ρυθμίσεις η Και πιστεύω ότι η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους. Εννοείται ότι μας ικανοποιεί το πρόγραμμα Leader και θα θέλαμε να επεκταθεί περισσότερο. Σε κάθε χώρα, σε κάθε κοινότητα θα θέλαμε να δούμε πολλές καλές πρωτοβουλίες. Για άλλη μια φορά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει περικοπή των κονδυλίων του Leader. Πάλι στο μισό περίπου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί το πρόγραμμα αυτό όχι μόνο ε, διατηρεί τη ζωή στις ε, περιφέρειες αυτές της υπαίθρου, διατηρεί τον κόσμο εκεί, τον κρατάει στα σπίτια του, στηρίζει επίσης τους νέους και τους ανθαρρύνει να μείνουν στην περιοχή. Φυσικά και γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες σήμερα. Από την άλλη θα θέλαμε περισσότερους νέους αγρότες να έχουν ευκαιρίες οι νέοι για να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο και να αναλάβουν εκεί δραστηριότητες. Επίσης, με την ανεργία που πλήττει τους νέους, Κάτω του 6% των αγροτών στην Ευρώπη είναι νέοι αγρότες. Χρειάζεται λοιπόν στήριξη στους νέους αγρότες, ακόμα περισσότεροι από αυτοί που έχουμε σήμερα, και να πούμε ότι η στήριξη αυτή θα δίνεται στους αγρότες μέχρι 45 ετών, όχι μέχρι 40 όπως προτείνεται, για να ενθαρρύνουμε περισσότερο κόσμο να αναλάβει δραστηριότητες στην Ήπεθρο, στη Γεωργία, να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις κλπ πρέπει επίσης να φροντίσουμε και την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό να το κάνουμε όχι μόνο με παραδοσιακές δραστηριότητες, αλλά να δούμε τι προπτικές υπάρχουν για το μέλλον. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφία στην Ήπεθρο. Χρειαζόμαστε όχι μόνο κερδοφόρο αγροτικό κλάδο, αλλά πρέπει να στηρίξουμε και τους τομείς εκείνους που είναι λιγότερο κερδοφόροι, αλλά που είναι πολύ βασικοί για τη διατήρηση της βιολογικής ε, ε, ποικιλομορφία ε, που κρατάει τον κόσμο στις χώρες του κτλ. 40% πρέπει να δίνεται στήριξη σε τομείς οι οποίοι είναι για το μέλλον, που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή μην ε, σταθούμε μόνο στα παραδοσιακά μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί στο μέλλον αυτά τα μέτρα, τα μη παραδοσιακά, θα φέρουν περισσότερα αποτελέσματα και θα είναι ένας υγιής ανταγωνισμός, όχι μόνο μεταξύ των χωρών μελών και των περιφερειών τους, Ξέρουμε ότι υπάρχει ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο που μερικές φορέ έχει αρνητικές συνέπειες ο ανταγωνισμό από τρίτε χώρες για παράδειγμα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό Εμεί να συνεχίσουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε τι υποχρεώσει μα. Τώρα όταν μιλάμε για την απλοποίηση πρέπει να πω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας, να περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, και να επιτρέπουμε στις χώρες μέλη να δημιουργούν τις δικές τους ε, ρήτρες ασφαλείας και επίσης να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μία λύση που να κάνει για όλους. Άρα να προσαρμόζουμε την πολιτική μας και να ε, αποθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να δημιουργούν τοπικά τη δικιά τους γραφειοκρατία. Κάτι άλλο, στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, είναι ότι πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια στους ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εδώ βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις όπου δεν προσφέρονται κοινωνικές εγγύησεις σε ανθρώπους που εξαρτώνται από την ε, γεωργία. Δευτερευόντως δηλαδή απασχολούνται στη γεωργία. Κάτι το οποίο τους δημιουργεί δυσκολίες βέβαια όταν δεν είναι ασφαλισμένοι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στο επίπεδο στήριξης. Μερικές φορές έχουμε διαφορές που είναι στο 1 τρίτο. Πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση, να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Το 2013 δεν κατάφεραν όλες οι χώρες να πετύχουν τον μέσο όρο. Και γι' αυτό θα έπρεπε να περιμένουμε την επόμενη περίοδο να μην έχουμε μόνο το 8%, να έχουμε πλήρη σύγκληση, 100% το 2027. Αυτό να προβλέψουμε. Και επίσης να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου σε κάποιες χώρες οι γεωργοί νιώθουν ότι είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Δεν έχουν ευκαιρίες εξαιτίας ακριβώς αυτών των διαφορών στα έσοδά τους. Ήδη σήμερα βλέπουμε δράσεις διαμαρτυρίας, διαδηλώσεις κάθε τόσο μπροστά στο κτίριο της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Την επόμενη εβδομάδα μάλιστα ή λίγο μετά, στις 13 Δεκεμβρίου, περιμένουμε μια νέα μεγάλη διαμαρτυρία επειδή και επιμένω ο κόσμος νιώθει ότι έχει το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες, σε ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες ανταγωνισμού. Και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Και έχουμε και σε ένα ακόμα θέμα που θέλω να καλύψω. Και εδώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λάθος. Πρόκειται για τους περιφερειακούς φορείς στην Ευρώπη. Από το 2016 βλέπουμε όλο και περισσότερες περιφέρειες να λειτουργούν από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν ε, έχει δεδομένα, αλλά στη χώρα μου, στην Τσεχία για παράδειγμα ή στη Λετωνία, έχουμε νέες περιφέρειες που δημιουργούνται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τις δέχεται, γιατί δεν έχει στατιστικά δεδομένα, λέει. Και τελικά θα βρεθούν σε μια κατάσταση το 2027 μόνο με τις περιφέρειες που υπήρχαν ήδη το 2016. Οι υπόλοιπε δεν θα καλύπτονται από το νομικό πλαίσιο. Μα είναι άδικο κάτι τέτοιο. Γιατί στις χώρες αυτές έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Ένα προς τέσσερα. Και γι' αυτό θέλουμε να μειώσουμε τις διαφορές. Να μειώνονται διαφορές δηλαδή στην Ευρώπη όχι μόνο μεταξύ των ε, διαφόρων χωρών μελών, αλλά μεταξύ και των περιφερειών. Υπάρχουν ε, τόσα χρήματα που δίνουμε, αλλά αν δεν ληφθούν υπόψη νέε περιφέρειες, κινδυνεύει το χάσμα να γίνει ακόμα μεγαλύτερο αντί να μειώνεται. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ήπεθρο. Γιατί ξέρουμε ότι ο πληθυσμός στην Ήπεθρο μειώνεται συνεχώς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί λείπουν υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες που επειδή δεν είναι οικονομικά αποδοτικές δεν προσφέρονται στην Ήπεθρο. Και το αποτέλεσμα είναι οι νέοι να φεύγουν. Ανακαλύπτουν την αδυναμία εφόσον ζουν σε τέτοιες περιοχές και φεύγουν και μετακινούνται στα αστικά κέντρα. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να το αντιστρέψουμε. Γιατί αλλιώ γίνεται χιονοστιβάδα. Αδειάζει η ύπεθρος, την εγκαταλείπει ο κόσμος, δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό εκεί, χέρια να δουλέψουν. Και αν όλα βασίζονται στην κερδοφορία, τότε προφανώς όλες αυτές οι υπηρεσίες δεν θα μπορούν να προσφέρονται, γιατί δεν είναι επικερδείς. Είναι όμως αναγκαίες για τον πληθυσμό, για την παραμονή του πληθυσμού εκεί. Σε αυτό λοιπόν θέλω να επιστήσω την ε, προσοχή σας. Και κάτι ακόμα, κάποιες ακόμα ιδέες θα σας πω για τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές ομάδες. Εάν υπάρχουν προγράμματα επιτυχή, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση που είχαμε και το, κατά το παρελθόν. Να μην γίνονται περικοπές σε αυτά τα επιτυχή προγράμματα. Αντίθετα, να δίνουμε την ευκαιρία στις τοπικές κοινότητες να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που έχουν. Να αποφύγουμε τις, τους ανοιχτούς διαγωνισμούς που βασίζονται μόνο στον ανταγωνισμό τον οικονομικό. Πολλές φορές βλέπουμε μια πρόταση με πολύ καλή περιγραφή, πολύ καλά στοιχεία. Στην πράξη όμως δεν είναι κάτι που ανήκει στην τοπική κοινότητα. Αν λοιπόν οι κεντρικές αρχές θέλουν λύσεις για τις τοπικές κοινότητες, γιατί να μην του δίνουμε προτεραιότητα. Τέλο πάντων, μπορεί να έχω μακρηγορήσει πολύ, θα σταματήσω τώρα, αλλά περιμένω τις δικέ σας προτάσεις και τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροπέ. Κύριος Πούτα δεν βλέπω να είναι εδώ, εκ μέρους του. Κυρία Καρσία Πέρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα εξήγησε εκτενώς ο εισηγητής ποια είναι η θέση του. Γενικά μιλώντας η αλήθεια είναι ότι στηρίζω περισσότερα από αυτά που είπε. Κάποιες παρατηρήσεις όμως έχω να κάνω κι εγώ. Πρώτον, πιστεύω ότι στην Επιτροπή μας θα έπρεπε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την πρόταση τη δημοσιονομική. Τα κονδύλια δηλαδή που διατίθενται στην αγροτική πολιτική. Το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί, είναι κατά των περικοπών στις παραδοσιακές πολιτικές, περιφερειακή, κοινή γεωργική πολιτική και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και καταλαβαίνουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι κάτι πολύ βασικό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεπώς, θα πρέπει να διατηρηθεί η θέση μας κατά των περικοπών γιατί η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει μείωση της τάξης του 15% για την περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι πολύ δυσάρεστο. Δεύτερον, με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποίησης της σημερινής κοινή γεωργικής πολιτικής γίνεται εισαγωγή νέων στρατηγικών σχεδίων έτσι όμως υπάρχει ένας κίνδυνος και το έχουμε πει αυτό πολλοί από εμά στην Επιτροπή για το ότι ο κίνδυνος είναι επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι κοινή και πρέπει να παραμείνει κοινή. Είναι πολύ βασικό αυτό για να μπορούμε να διαχειριστούμε την επικράτειά μας. Οπότε και αυτό πρέπει να το προσθέσουμε. Και τώρα έρχομαι στα βασικά που έχουν να κάνουν με τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση των στρατηγικών αυτών σχεδίων. Αναφερθήκατε στο θέμα της γυναίκας. Ε, αυτό ε, εγώ θέλω να το βάλω σε ένα ψηλό επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να ενσωματώσουμε και ένα νέο στόχο σε αυτούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μιλάει για τα έσοδα, για τις αγορές, για τους νέους, για το περιβάλλον τέτοιου στόχου. Ωραία, όλοι αυτοί οι στόχοι είναι καλοί, αλλά νομίζω ότι στο ίδιο επίπεδο πρέπει να μπει και ο στόχο των ε, δικαιωμάτων τη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα πάντα ήταν βασικό στοιχείο στην ε, διατήρηση της υπαίθρου και θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο το έργο των γυναικών στην υπαίθρο. Πρέπει λοιπόν στη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής να συμπεριλάβουμε και συγκεκριμένα στοιχεία πάνω σε αυτό. Επίσης πρέπει να συμπεριλάβουμε στους στόχους αυτούς και το ζήτημα που έχει να κάνει με τη διατήρηση του πληθυσμού. Η Επιτροπή μας και ολόκληρο το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε με έκθεση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία και μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας, την ΚΑΠ για παράδειγμα, για να διατηρηθεί ο κόσμος στην Ήπεθρο. Τα στρατηγικά μας σχέδια λοιπόν πρέπει να προβλέπουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση ε, της απερίμωσης της υπέθρου για να δημιουργείται απασχόληση εκεί, να αποτελεί σε ελκυστικό χώρο που να δίνει δυνατότητες για την εγκατάσταση νέων, για δραστηριότητες, κυρίως για νέους και για γυναίκες που να μπορούν στην Ήπεθρο με τα μέτρα αυτά να ε, δημιουργήσουν επιχειρήσεις, μια νέα δραστηριότητα, πας περιπτώσει. Και τελειώνω με δύο στοιχεία ακόμα, πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, για τη σύγκληση. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο συγκητής. Όντως, πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της εξωτερικής σύγκλησης. Αλλά θεωρώ ότι το να το κάνουμε αυτό, αυτή την περίοδο, σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο. Γιατί λέμε ότι έχουμε λιγότερα χρήματα για την ΚΑΠ και να κάνουμε εξωτερική σύγκληση σε λίγο χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει η οικονομική διόρθωση. Πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί έτσι θα υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση της ενίσχυσης. Οπότε συμφωνώ με το στόχο της εξωτερικής σύγκλησης, αλλά πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσαρμοστούμε σε αυτό με το χρόνο. Επί της αρχής συμφωνώ. Και τέλος, κάτι επίσης συγκεκριμένο, που είναι σημαντικό για την περιφερειακή πολιτική. Το θέμα των μόνιμων λιβαδιών. Θυμόσαστε ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε συζητήσει πολύ ε, για το πώς θα ορίσουμε τι είναι αυτό. Γιατί για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας, της κτηνοτροφίας κυρίως, είναι πολύ σημαντικό για κάποιες περιοχές και υπήρξαν ε, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και τις χώρες μέλη. Σε αυτή την νέα μεταρρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι εξαφανίζεται ο ορισμός ο οποίος είχε συμφωνηθεί, ενώ είχαμε συμφωνήσει όλοι. Θα πρέπει να επανέλθει αυτός ο ορισμός που είχαμε εγκρίνει στον κανονισμό Omnibus για το τι είναι τα μόνιμα λιβάδια. Στο περιφερειακό τομέα είναι πολύ βασικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για το έργο του και εννοείται ότι είμαι και εγώ ε, στην διάθεσή του να συζητήσουμε όταν έχουμε τροπολογίες ευχαρίστως για να ετοιμάσουμε ένα κείμενο πάνω στο οποίο θα υπάρξει συνένεση μεταξύ όλων και θα καλύπτονται όλες οι θέσεις. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα αυτό η εδώ. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να παρουσιάσω εγώ την ε, τοποθέτηση της κυρίας Κάτα. Είναι ένα εκ μέρους της Άλτε που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Με παρακάλεσε λοιπόν να κάνω ανάγνωση της θέσης της. Η κυρία Κάταινεν θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τις πολλές αξιόλογες ιδέες του σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική και σχέδιο, την πρόταση για το στρατηγικό σχέδιο. Είναι εν γέννη σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο ευελίξης για τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τα εθνικά σχέδια, αφού η γεωργία και ο γεωργικό τομέα οι διάφοροι τομεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Γεωργίας παρουσιάζουν ποικιλομορφία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους τη δυνατότητα να εξειδικευθούν στα ε, οικεία, με βάση τα οικεία ε, σχέδια κουγουπού, να ενισχυθεί η εθνική πολιτική, να ενισχυθεί η επικουρικότητα σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προτάσεις για βελτίωση της περιφερειακή ανάπτυξη και διάφορες ιδέες που έχουν σημασία για την ε, οπτική της Επιτροπής μας είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν όχι μόνο οι αρχικές φάσεις των γεωργικών επιχειρήσεων, των νεοφιών επιχειρήσεων όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η περαιτέρω εξέλιξη φυσταμένων μικρό και μικρότερων επιχειρήσεων στην Ήπεθρο. Πρέπει επιπλέον να εξασφαλιστεί ένα ευρύ φάσμα ε, επιχειρήσεων στην Ήπεθρο, η νεοφύης και η ανάπτυξη της βιολογικής οικονομίας, της κυκλικής οικονομίας, της, του τουρισμού αλλά και άλλων τομέων δραστηριότητες. Το άρθρο 69 και η επίκλησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περιορισμένο φάσμα ως εκ τούτου και αναφέρεται μόνο στη γεωργία και τη δασοπονία που μπορεί να είναι σημαντική το τομή, ωστόσο θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση. Η τωρινή πρόταση θα απέκλεινε δηλαδή όπως έχει στο μέλλον επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ζωτική σημασία για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, η αναπτυξιακή βοήθεια έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ε, δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιβίωση και μη γεωργικού χαρακτήρα επιχειρήσεων και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ως πολύ σημαντικό. Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση της κυρίας Κατάινεν. Ο κύριος, η κυρία Ντεμάτου δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ τους λοιπούς συναδέλφους που ε, επιθυμούν να τοποθετηθούν με τον κύριο Πόλτσεκ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί η ΚΑΠ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι κλιματολογικές αλλαγές σε πολλούς τομείς, όπως το εμπόριο. Είναι απαραίτητο επίσης να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της κυκλικής οικονομίας. Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα, είναι θα έλεγα απαραίτητο αυτό για τη γεωργία και ιδιαίτερα για τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αντίθετα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές γενικά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, μειονεκτούν Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τα προβλήματα της ποιότητας της γης. Αν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει σήμερα, ε, τότε φοβάμαι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα είναι ακόμα ισχυρότερες και οι μικρές ακόμα θα γίνουν ασθενέστερες. Σχετικά τώρα με το ΦΕΝΤΕΡ, νομίζω ότι όχι μόνο δεν θα πρέπει να μειωθεί, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν τρόποι αύξησης του συνολικού πακέτου. Θα πρέπει επίσης το κομμάτι του Ταμείου Εγγυήσεων και του Λίντερ να αυξηθούν σημαντικά. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές να λειτουργήσουν λοιπόν με σωστό τρόπο και να χρησιμοποιήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο τις δυνατότητες επένδυσης στις γεωργικές περιοχές. Θα συμφωνήσω επίσης μαζί σας και σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς όπως το ΦΕΟΓΑ, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους νέους και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. θα βοηθήσει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. οι επιδοτήσεις, η βοήθεια μάλλον γενικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μερικές φορές δεν καταλήγει εκεί που πρέπει. Εποφελούνται μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κάνουν περίεργες δηλώσεις και διαιρέσεις σε σχέση με το μέγεθός τους. Το θέμα αυτό είναι θέμα φυσικά ελέγχου, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πράγματι τίθεται. Πρέπει όλα αυτά λοιπόν να τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Ευχαριστώ κύριος Μπόγκοβιτς. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Η κοινή αγροτική πολιτική βασίζεται ουσιαστικά στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σαν στόχο να διασφαλίσει επαρκείς ε, συνθήκες ζωής στους αγρότες. Αν αναλύσει κανείς τις νέες προτάσεις και τον ρόλο τον οποίο ε, μπορεί να παίξει η κοινή αγροτική πολιτική, Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς είναι πάρα πολλές. Έχουμε προβλήματα ήδη και στον τομέα της σύγκλησης. Έχουμε θέματα σε σχέση με τη δίκαιη κατανομή ανάμεσα στις χώρες μέλη. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές οι οποίες δεν δείχνουν να μειώνονται. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά στάσεις συγκέντρωσης των εδαφών. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι όλοι όσοι ωφελούνται από τις δυνατότητες που παρέχονται το αξίζουν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις δυνατότητες που ε, παρέχει η επικουρικότητα. Έχουμε ένα πλαίσιο, ένα κανονισμό πλαίσιο και αυτό είναι σχετικά καινούριο έρχεται από τις συνθήκες βέβαια, προβλέπεται από τις συνθήκες Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η ΚΑΠ έτσι όπως λειτουργεί σήμερα δεν είναι ικανοποιητική. Και όλα τα ποσά τα οποία είναι διαθέσιμα για τη συνοχή τείνουν να μειούνται, ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να ισχύει. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε με μεγαλύτερες ευθύνες τα κράτη-μέλη. Από ό,τι φαίνεται ότι έτσι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να, συνεχώς, να παραπονούνται συνεχώς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά υπάρχει παρόλα αυτά ένας κάποιος κίνδυνος εδώ. και θα είναι δύσκολο να θέσουμε σε λειτουργία κάποια στρατηγικά θα έλεγα προγράμματα κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Αυτά θα τα δούμε πάλι στις επόμενες συζητήσεις. Προτείνω σαν παράδειγμα την παράταση ε, της ε, μεταβατικής περίοδου και θα πρέπει να ωφεληθούμε επίσης από αυτούς οι οποίοι είναι δραστήριοι στον τομέα αυτό εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τα ποσά αυτά έτσι ώστε και οι λιγότερο νέοι να μπορέσουν να ωφεληθούν. Αυτά συνδέονται γενικότερα με την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης, όπως επίσης και με το πρόγραμμα Τα Leader. Και δεν καλύπτουμε εδώ μόνο τους γεωργούς. Θα πρέπει να επενδύσουμε επίσης στις υπηρεσίες υγείας, στην έρευνα, και νομίζω ότι η πρωτοβουλία για το FES χωριό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε τους ίδιους στόχους. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να δώσουμε σε αυτήν την εκστρατεία μια νέα ζωτικότητα. Ελπίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να δημιουργήσουν νέους μηχανισμούς, μηχανισμούς απαραίτητους έτσι ώστε να προωθήσουμε τις πολιτικές που έχουμε αποφασίσει. Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Έχω δύο παρατηρήσεις. Στην περιφερειακή πολιτική έχουμε δουλέψει πολύ για την ευφύη δίκευση. Οι χώρες μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δούμε πού είναι η δύναμή τους και σε αυτή να μιζάρουμε. Άλλος είναι στην ψηφιακή οικονομία, Εξαρτάται δηλαδή σε τι είναι καλό η κάθε περιφέρεια. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι το θέμα δεν είναι τόσο για τη γεωργία και τα προϊόντα, είναι και μετά για την επεξεργασία. Δηλαδή, αν κάποιος παράγει και η αγορά δεν παίρνει, πρέπει να κάνουμε αυτήν τη σύνδεση ακριβώς. η γεωργική παραγωγή δεν είναι μόνο τρόφιμο, είναι και πρώτη για την ε, κυκλική οικονομία. Δηλαδή ο σπόρος ε, μπορεί να συγκριθεί με την ε, ορυκτήλη. Οπότε λοιπόν εδώ θα ήθελα να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τις παλιές χώρες μέλη που τεχνολογικά μπορεί να έχουν προωθηθεί περισσότερο, που αποτελούν ένα πόλο ανάπτυξης, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες χώρες από, και οι περιοχές από όπου φεύγει ο κόσμος. Αυτή η ευφύης δίκευση είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθεί έτσι κάποιο οικοσύστημα και να είναι κάτι ελκυστικό, δηλαδή να μπορούν να πηγαίνουν νέες επιχειρήσεις και να συνεργάζονται με τους αγρότες με μια μορφή συνεταιριστική ίσως. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Δεύτερον, για την κοινωνική πτυχή. Ναι, λέμε ότι σε πολλές περιφέρειες έχει φύγει ο μισός πληθυσμός. Στην Ανατολική Πολωνία, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι. Και είχαμε και το ψήφισμα που εγκρίναμε πριν από δύο λομέλειες ακριβώς ώστε η νέα τεχνολογία, η γνώση να φτάσει παντού και να εξυπηρετήσει όλες τις περιφέρειες. Πρέπει να σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων που έχουμε τελευταία και στην Ευρώπη. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Και αυτή ήταν η τελευταία τοποθέτηση από τους ε, βουλευτές της Ρέτζη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μπορεί να λάβει το λόγο. Ο κύριος Μιλούσεφ από τη βλέπω στις μειώσεις μου θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, εξωτικό μέλη της Επιτροπής. Αναφέρθηκαν οι περισσότεροι ομιλητέ στον προπολογισμό, για να μην πω όλοι. Και ξεκινώ από αυτό λοιπόν. Βεβαίω, η περιφερειακή ανάπτυξη επιτυχή θα είναι όταν θα έχουμε επαρκεί πιστώσει. Ωστόσο, θα πρέπει και να αναγνωρίσουμε ότι η δράση μας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο που καθίσεται ακόμα πιο περίπλοκη λόγω του Brexit. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτονται στο νέο πλαίσιο νέες προτεραιότητες όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση. Και έτσι έχουμε αυτούς τους περιορισμούς. Από την άλλη, μέσα σε αυτά τα όρια πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή υποστήριξη για τις περιοχές της Υπέθρου. Η ΔΕ Επιτροπή έχει δηλώσει απερίφραστο ότι δεν σκοπεύει να περικόψει την υποστήριξη. Απλώς θέλει να εξισορροπήσει τις δαπάνες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και στοχεύει σε, επιδιώκει καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν, συνεργατικές σχέσεις, συνεργασίες με άλλα μέσα χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, και άλλα νομοθετήματα θα είναι πάντα χρήσιμες. Επίσης υπογραμμίζω την δυνατότητα για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των πυλώνων, δηλαδή πέραν της συνήθους ε, μεταφοράς έχουμε τη δυνατότητα για 15% αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε άλλο ένα 15% ε, δυνατότητας μεταφοράς από την περιφερειακή ανάπτυξη στο περιβάλλον χωρίς ε, πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση. Επιπλέον αυτού στον πρώτο έχουμε τη δυνατότητα για υποχρεωτικό οικολογικό πρόγραμμα που είναι ένα μέτρο ισοδύναμο θα προς την περιφερειακή ανάπτυξη και επιτρέπει εκεί πέρα την ενίσχυση των δαπανών. Και επίσης, για να απαντήσω και σε κάποιες άλλες παρατηρήσει που διατυπώθηκαν, ξεκινώντας με το Leader, ε, ακούστηκε ότι το Leader έχει περικοπεί κατά δύο μισή φορές. Δεν βλέπω από πού ε, αντλείται αυτή η πληροφορία του εναντίον. Εμείς έχουμε ε, Έχουμε επιβάλει την υποχρέωση για διατήρηση κατά 5% του Λίντερ και αυτό λόγω της εμπειρίας που έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να προχωρήσουν ακόμη και παραπέρα. Μένει το 10%. Έχουμε και κράτη όπου σε περιφερειακούς όρους το Λίντερ έχει φτάσει και στο 30%. Αυτές τις δυνατότητες τις διατηρούμε. Και θα είναι ακόμη λιγότερο ε, γραφειοκρατικό στο μέλλον. Θα ένα πλαίσιο συνεργασίας, ένα μέτρο συνεργασίας με μεγάλο βαθμό ευελιξίας γιατί προσφέρει και περισσότερες δυνατότητες δράσης των τοπικών ε, κοινοτήτων και επιλογών. Μια άλλη παρατήρηση για τους νέους γεωργούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αυτούς, προτεραιότητα άλλωστε αποτελούν οι νέοι γεωργοί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον με ένα 2% τουλάχιστον των πιστώσεων από τον πρώτο πυλώνα σε όρους ισοδυνάμου και επίσης το όριο ηλικία λένε κάποιοι να ξεπεράσει τα 40 έτη. Δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Θα είναι λιγότερο στοχευμένη τότε η στήριξη που θα μπορούμε να προσφέρουμε και έχοντας κάνει τη σχετική μελέτη αλλά και εμπειρία θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουμε ε, σε συγκεκριμένους στόχους και άρα στα 40 έτη ηλικίας. Βέβαια καθής μπορεί να ε, συζητεί το τι σημαίνει νέο στη σημερινή μέρα, αλλά για μας όριο θα είναι τα 40. Επίσης πρόταση για την κλιματική αλλαγή. Να πάει αυτή στα 30%. Έστω αλλά στην κοινή γεωργική πολιτική ο προϋπολογισμός ε, και η ε, προσδοκία για συμμετοχή τους στις κλιματικές Στου κλιματικούς στόχους θα είναι στο 40%. Επομένω αντίστοιχα, περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υποστήριξη αυτών των επιλογών για την κλιματική πολιτική. Για τους άλλους γεωργού περιορισμοί δεν υπάρχουν ε, εάν ανταποκριθούν, δηλαδή αν ανταποκρίνονται στα κριτήρια χρηματοδότηση νέοι ε, ε, γεωργοί δεν έχουν περιορισμούς, είτε προέρχονται από το αστικό κέντρο είτε από την Ήπεθρο. Σύγκληση, ε, ακούστηκαν δύο διαφορετικές απόψεις σήμερα. Η πρώτη του κυρίου Ροπέ που μας λέει ότι θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε την εξωτερική σύγκληση μέχρι το τέλος της προγραμματικής περίοδου. Αλλά υπήρξε και η αντίδραση της κυρίας Γκαρσία Πέρες που είπε ότι δεν είναι σωστό αυτό σαν επιλογή. Το ίδιο βλέπουμε όμως και από το Συμβούλιο. Άλλα κράτη-μέλη ζητούν περισσότεροι, άλλοι λιγότεροι και εμει καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δική μας πρόταση είναι καλή και λογική. Τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν μείωση σε 3,9% των ε, αμεσών ενισχύσεων εφόσον το επιλέξουν σε επίπεδο αναεκτάριο κάτω από αυτό το οποίο ορίζεται σε εθνικό μέσο όρο μπορούμε να έχουμε αύξηση ε, μέχρι 4%. Ας μην το λησμονούμε λοιπόν αυτό, ότι υπάρχει δυνατότητα και για διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Στο επίπεδο αναγνωρίσεως τώρα των ε, περιφερειών πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ της γεωργικής και της περιφερειακής πολιτικής για να υλοποιούνται καλύτερες στόχοι, κοινωνικές πτυχές που ανέφεραν αρκετοί ομιλητές, κοινωνική στόχοι, κοινωνική γεωργία. Αυτό που ήθελα να φέρω εγώ είναι ότι έχουμε στον κανονισμό, στο άρθρο 3, ε, τρεις στόχους συγκεκριμένους που θεωρούμε ότι επαρκούν για να καλυφθεί το σύνολο των προκλήσεων που αναφέρθηκαν άλλωστε και εδώ, περιφέρεια δηλαδή, ύπεθρος μάλλον, γυναίκες, κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται να ε, συμπληρώσουμε με περισσότερους στόχους. Σημαντικό θα είναι αυτά που θα σχεδιάσουν τα κράτη-μέλη να είναι καλές επιλογές. Αυτό λοιπόν το υποστηρίζουμε, απλώς επισημαίνω ότι δεν πρέπει να παραφορτωθεί ο κανονισμός με πληθώρα στόχων και επαναλαμβάνω θα κρυθούν τα πάντα από τα όσα θα ε, περιλάβουν στα προγράμματά τους τα κράτη-μέλη. Περιορισμούς όμως πρακτικά δεν έχουμε επιβάλει. Και συνεχίζω. Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν οπισθοδρομούμε. Εδώ αυτό θα απαντήσω μόνο. Αυτό που κάνουμε είναι ότι στρέφουμε το βλέμμα προς τον μέλλον και δίνουμε δυνατότητες για το γενικό πληθυσμό μέσω του κανονισμού που μπορεί να επιλέξει το κράτος μέλος. Άρθρο 69. Ε, επιχειρήσεις της υπαίθρου και μη ε, γεωργικές επιχειρήσεις της υπαίθρου. Αντιλαμβάνομαι τα επιχειρηματά σας, αλλά εδώ έχουμε δύο πολιτικές. Και, τη, και την συνοχή η περιφερειακή πολιτική, αλλά και την γεωργία αφετέρου. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ε, κάποιος διαχωρισμός, κάποιο όριο μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών. Έχουμε επιβάλει αυτούς τους ε, περιορισμούς στις προτάσεις μας. Επίσης και καθώς υπήρξαν διάφορες ε, παρεμβάσεις, θα ήθελα να επισημάνω για να λάβετε υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά πολλά χρόνια που η βιοοικονομία και οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής συντονίζονται και Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά ε, για την κυκλική οικονομία, εξειδικεύση των αγορών κτλ. Όχι μόνο μέσω της ΚΑΠ, αλλά και γιατί υπάρχουν δυνατότητε δυνατότητες και από την κυνηγιορική πολιτική βεβαίως και από την ΚΑΠ, αλλά και γιατί τα ποσά που προβλέπουμε στον ορίζοντα 2020 ε, διπλασιάζονται με τον προϋπολογισμό αυτών και δίνουν έτσι νέες δυνατότητες στον τομέα αυτών. Δεν ξέρω αν έχω καλύψει όλες τις παρατηρήσεις, μάλλον όχι, αλλά θα σταθώ σε αυτά τα σχόλια και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σημειώσω ότι έχουμε ένα νέο μοντέλο οικονομίας. Α, όχι, πολύ σημαντικό ήταν αυτό που είπε η κυρία Γκαρσία. για την ανανέωση των νέων έχει απαντήσει ο, ο Επίτροπος, διαφυλάσσουμε το επίπεδο, διαφυλάσσουμε... Εμείς ορίζουμε τους δείκτες ε, σύμφωνα με την βάση εκπλήρωσης του στόχου. Εκεί υπάρχει περισσότερη επικουρικότητα, όχι στην πολιτική τη δική μας, αλλά στην εφαρμογή της πολιτικής. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια του νέου αυτού πακέτου, του νέου αυτού μοντέλου αν θέλετε παροχής ε, των συγκεκριμένων προγραμμάτων έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Φυσικά εμείς δεν είμαστε εναντίον της αύξησης στον προϋπολογισμό αν αυτό είναι κάτι το εφικτό. Λοιπόν, 29 Νοεμβρίου 12η μεσημβρινή προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Κύριε Ροπέ, θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Νομίζω ότι ήταν ζωηρή η συζήτηση, χρήσιμη συνεπώς. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και τις ιδέες σας. Εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, υπήρξαν και κάποιες επικαλύψεις. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναζητήσουμε λύσεις και στις δύσκολες ε, ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική και τα στρατηγικά προγράμματα υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει κανείς με 27 διαφορετικές γεωργικές πολιτικές. Γι' αυτό απαιτούνται ορισμένες ρήτρες ασφαλείας για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αν τώρα τα κράτη-μέλη αρχίσουν να κάνουν αποκλίνουσες δικές τους πολιτικές, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση και το επίπεδο ανάπτυξης ανάμεσα στα κράτη-μέλη θα αρχίσει να διαφέρει ε, ακόμα περισσότερο. Σχετικά με τη σύγκληση, έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου οι προσπάθειες για τη σύγκληση πρέπει να καρποφορήσουν επιτέλους. 20 χρόνια έχει κρατήσει ε, οι προσπάθειες αυτές. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει με το ζόρι να παίρνουμε λεφτά από τη μία χώρα και να τα δίνουμε στην άλλη αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν δυνατότητες έβρεσης επιπλέον χρηματοδότησης εκεί όπου χρειάζεται. Οι προτάσεις που έγιναν σχετικά με τα μέτρα αναζωογόνησης της υπαίθρου μου αρέσουν πολύ. Και με τη στήριξή σας τα μέτρα αυτά θα τα προωθήσω και θα τα καταθέσω. Είναι δυνατόν να είμαστε εφάνταστοι και καινοτόμοι ηλεκτρονικό εμπόριο, βιοτεχνικές δραστηριότητες ε, με βάση την τοπική παραγωγή σε τοπικό επίπεδο και με τοπικά προϊόντα. Σαν παράδειγμα τα υποπροϊόντα της δασοκομείας. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε οι τοπικοί πληθυσμοί να βρίσκουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται ε, και τοπικά προϊόντα και στις τοπικές αγορές και σε καλές τιμές. Πρέπει να επιλέξουμε όλοι ε, το πρότυπο της ε, μικρής αλυσίδας, δηλαδή να στηρίζουμε τις τοπικές υπηρεσίες και, τις τοπικές, και τα τοπικά προϊόντα. Έτσι θα μπορέσουμε νομίζω να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε τη ζήτηση που τόσο λείπει ε, στις ε, αγροτικές περιφέρειες. Και η ύπεθρος δεν θα πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά ε, στα προϊόντα τα γεωργικά, αλλά να συνδυάζει τα προϊόντα αυτά και τη γεωργία γενικότερα με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και έτσι θα φέρουμε και πιο κοντά τις αστικές περιοχές με τις περιοχές της υπαίθρου καθαρού γεωργικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Thank you very much. So... Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία λοιπόν 29 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι. Θα συνεχίσουμε τώρα με το γεωργικό τομέα πάντα. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση. Η υπεύθυνη επιτροπή είναι η Άγκρη. Έχουμε προετοιμάσει μια ε, ε, γνωμοδότηση. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στην έκθεση αυτή στη στρατηγική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε και αναφέρομαι εδώ και στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εν πολλής ε, θα έλεγα ότι είναι επαναστατική. Η πρόταση αυτή δημιουργεί ουσιαστικά τις δυνατότητες ουσιαστικής μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής την εξυγχρονίζει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές στο μέλλον. Ποια είναι η βασική αλλαγή, η σύγκληση καταρχάς. Η σύγκληση η οποία μέχρι τώρα γινόταν αντικείμενο διαχείρισης από τις Βρυξέλλες, τώρα στην ουσία μετατρέπεται σε παρακολούθηση των επιδόσεων και ε, με πολύ στοχευμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους περισσότερη ευελιξία, περισσότερη επικουρικότητα και κυρίως αυτήν την ευελιξία μπορεί να την ε, οδηγήσουν στην προσπάθεια μείωσης των διαφορών ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές στον τομέα αυτό, ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές ευθύνες, διαφορετικές ε, προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα για την αξιολόγηση και την εποπτεία των επιδόσεων και των δικτών με βάση τους δείκτες τους οποίους χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, ε, σε σχέση δηλαδή με το τι παρακολουθούμε και ελέγχουμε και τι αφήνουμε εκτός ελέγχου. Συνεπώς θα περάσουμε σε μικρότερα γραφειοκρατικά βάρη, θα περάσουμε σε απλούστευση των διαδικασιών και θα έχουμε γενικά ένα νέο πρότυπο παρέμβασης. Ξέρετε ότι ο τέος πρώτος πυλώνας και ο δεύτερος τώρα συνδυάζονται μέσα στο νέο κανονισμό ο οποίος γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν σε εθνικό επίπεδο. Διερωτώ αν η απλούστευση αυτή ε, φαίνεται εύκολα στη συγκεκριμένη πρόταση. Μήπως ε, η απλούστευση αυτή στην ουσία ε, σε μία πρώτη φάση τουλάχιστον αυξήσει για τα κράτη-μέλη τις γραφειοκρατικές δυσκολίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει λιγότερος έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχουν μικρότερες ε, λογιστικές διαδικασίες ελέγχου από τις διάφορες υπηρεσίες που εξαρτώνται από τις Βρυξέλλες. Γιατί να μην χρησιμοποιούμε το δίκτυο το δορυφορικό το οποίο υπάρχει σήμερα. Είναι μια επιπλέον επιλογή. Ξέρω ότι υπάρχουν εδώ κάποια ερωτηματικά και κάποια από τα στρατηγικά αυτά προγράμματα από ό,τι φαίνεται δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρα. Συνεπώς, ε, με βάση λοιπόν τον κανονισμό αυτό μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στον κανονισμό CMO για να συνδυάσουμε καλύτερα το σύνολο των στόχων και να συντονίσουμε καλύτερα τον σύνολο των στόχων. Αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα είναι να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα και αυτό περιλαμβάνεται και στον κανονισμό Omnibus. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και την εξωτερική και την εσωτερική σύγκληση και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά έχει διαμορφώσει κάποιους καλούς στόχους Ξέρω ότι ε, γίνονται τεράστιες αλλαγές ε, στις διάφορες χώρες στον τομέα αυτό και οι συνέπειες τους ε, θα πρέπει να ελεγχθούν και θα πρέπει να περιοριστούν. Λοιπόν, Το κάπινγκ ας πούμε τα ανώτατα όρια δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να είναι τα ίδια ε, σε ε, όλες τις χώρες ή σε κάποιες χώρες θα υπάρχουν διαφορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να βρούμε κάποιες λύσεις. Χθε όλα αυτά άλλωστε ήταν αντικείμενο συζήτηση και στην Επιτροπή Γεωργίας. Το θέμα είναι πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις αυτές έτσι ώστε να προωθήσουμε ένα πιο, ε, μια πιο δραστήρια ύπεθρο από ό,τι στο παρελθόν και όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχουν εδώ πολλές πολιτικές, η πολιτική σύγκληση, η γεωργική πολιτική και η περιφερειακή πολιτική. Και οι τρεις αυτές πολιτικές θα πρέπει να συνδυασμούν έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του τομέα και θα καλύψουν εν μέρη και το θέμα των μεταναστευτικών ρευμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να φαίνονται πλέον και στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης και μην ξεχνώντας εδώ και τον ρόλο τον πολύ σημαντικό του Κοινωνικού Ταμείου. Υπάρχουν επιμέρους προγράμματα για συγκεκριμένους τομείς όπως το Horizon, το Erasmus κτλ. Αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνουμε έξω τη λογική, την διάσταση μάλλον, της ανάπτυξης της υπαίθρου. Θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους την απερίμωση του πληθυσμού και θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους και τη φυγή ε, των πολιτών από τις φτωχότερες προς τις πλουσιότερες χώρες. Απαιτείται περισσότερη επικουρικότητα, απαιτείται περισσότερη απλοποίηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες τους και όχι να τα περιμένουν από τις Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να λειτουργήσουν με πιο εφάνταστο τρόπο εφόσον έχουν αναλάβει περισσότερες ευθύνες από ό,τι στο παρελθόν και στη συνοχή. Έχουν επιδείξει στο παρελθόν ότι είναι σε θέση να φανούν, να φανούν δημιουργικά τα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί οι οποίοι να έχουν σαν στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων γιατί οι καθυστερήσεις και στον τομέα της συνοχής και στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου δυστυχώς προκαλούν τρομακτικές συνέπειες. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπάρχουν άλλες τέτοιου είδους όπως το παρελθόν καθυστερήσεις. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η αρχιτεκτονική των δύο πυλώνων της κοινή αγροτικής πολιτικής Είναι κάτι το οποίο έχει μια κάποια αξία. Δεν χρειάζεται εμεί να τροποποιήσουμε το σύνολο του συστήματος γιατί έχει αποδώσει αρκετά. Τώρα για τους δείκτες σε σχέση με τον υπολογισμό της ετήσιας επίδοσης και τα λοιπά, εδώ υπάρχουν ίσως διάφορα επιμέρους θέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν πιο ξεκάθαρα. Να έλθω τώρα στις τροπολογίες. Το Κοινοβούλιο έχω την εντύπωση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αναλάβει ένα υψηλότερο επίπεδου ρόλο. Όλες ε, αυτές οι προβλέψεις ε, θα πρέπει ε, να ρυθμίζονται και μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο στον τομέα της εφαρμογής. Λοιπόν, λιγότερες εφαρμοστικές πράξεις, περισσότερες κατεξουσιοδότηση πράξεις, έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να προωθήσει την άποψή του. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η κοινή αγροτική πολιτική στην ουσία θα απεισχναθεί και θα καταστεί, θα καταστεί στο μέλλον μια αυστηρά εθνική πολιτική. Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες κατουσιοδότηση πράξεις. Στα πλαίσια της εφαρμογής λοιπόν της πολιτικής αυτής θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίσει εκ των έσω το τι συμβαίνει επί τόπου στις ε, διάφορες περιοχές της Υπέθρο. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε και πέρυσι με τη διαδικασία του Omnibus. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Το 2021 νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ρεαλιστική ημερομηνία. Εγώ προτείνω μια μεταβατική περίοδο διατούς, διετούς διάρκειας. Έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, τους μηχανισμούς και τα συστήματα, τα πληροφορικά, τα οποία θα μπορέσουν να προωθήσουν τις πολιτικές. Από το 21 και μετά λοιπόν διετής μεταβατική περίοδος. Σχετικά με την περιγραφή, την αναφορά που θα ε, χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των περιπτώσεων, όχι 15 Φεβρουαρίου, 15 Απριλίου σε αιτήσια βάση. Αν πράγματι θέλουμε οι εκθέσεις αυτές να είναι ποιοτικές σχετικά τώρα με τις αποκλήσεις. Οι αποκλήσεις ε, που οφείλονται ίσως σε ανώτερη βία, στον θάνατο ή στην αναπηρία ε, του συγκεκριμένου αγρότη κτλ. Κάποιες φορές ε, ορισμένες φυσικές καταστροφές είναι έτσι και λιώς αδιαφυσβήτητα μια ανώτερη βία και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε στην περίπτωση έκδοσης ε, αποκλήσεων, αδειοδότησης αποκλήσεων. Αλλά αν έχουμε ας πούμε 7 εκατομμύρια δικαιούχους δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους 100 δικαιούχους οι οποίοι την χάνουν μιας κάποιας εξαίρεσης απόκλησης. Το σύστημα λοιπόν δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει. Μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το copy-paste και να προσπαθήσουμε να περάσουμε στον καινούριο κανονισμό τον παλαιό και να μην επιβαρύνουμε με πολλή γραφειοκρατία τους μικρομεσαίους. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι έχουμε όλο το σύστημα της αγροτικής πολιτικής. Η Σκιώδης τώρα, η κυρία Γκαρθία πρώτα απ' όλα, αλλά σας παρακαλώ πολύ να είσαστε σύντομοι. Μην ανησυχείτε, ναι. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομη, ενώ οι συνόδελφοι μπορούν να μακρηγορήσουν περισσότερο. Λοιπόν, πρώτον, ένα θέμα που είναι σημαντικό και είναι αναγκαίο είναι να ανακτήσουμε το μηχανισμό αντιστάθμισης πόρων εφόσον ε, επιστραφούν ε, χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να είχαν δοθεί. Άπαξ λοιπόν έχει πληρώσει κάποιος περισσότερο ή λιγότερο, τον επόμενο χρόνο μπορεί να γίνει αυτή η αντιστάθμιση με την αντίστοιχη πληρωμή, να μην χρειάζεται να περιμένουμε χρόνια για να γίνει αυτή η διόρθωση. Νομίζω ότι είναι εύκολο να επαναφέρουμε δηλαδή το μηχανισμό αντιστάθμισης. Δεύτερον, με την ε, τωρινή μεταρρύθμιση, τα στρατηγικά σχέδια κτλ. Θα υπάρχουν ε, χώρες που ανάλογα με το εδαφικό θα έχουν ε, περισσότερους από έναν οργανισμό πιστοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ένας οργανισμός θα συντονίζει όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή όταν υπάρχουν αναπεριφέρεια ε, διαφορετικοί ε, συντονιστικοί οργανισμοί πιστοποίησης, να υπάρχει ένας ο οποίος θα συντονίζει όλους τους επιμέρους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ραπέ, παρακαλώ να είστε σίγουροι. Ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η γεωργική πολιτική, αλλά παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε, για τη γνωμοδότηση. Πολλά μου αρέσουν σε αυτήν. Και έχω όμως κάποιες τροπολογίες που θα υποβάλω έγκαιρα. Πράγματι, ήσασταν σύντομο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια από τους συναδέρφους. Όχι. Ωραία. Οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπόσμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη δράσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντω ήταν πολύ Ενδιαφέρονται όλα όσα άκουσα και εδώ στην Επιτροπή σας και στην Επιτροπή Γεωργίας. Τώρα για τον οριζόντιο κανονισμό συγκεκριμένα θα περιοριστώ να αντιδράσω στα σχόλια του συντάκτη στις τροπολογίες και σε αυτά που είπε η κυρία Πέρες. Πρώτα απ' όλα, για την μεταβατική διευθέτηση. Ξέρετε ότι ήταν πολύ νωρίς το 2021. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια πάντα έχει μεταβατικές διευθετήσεις, συζητήθηκε με τις χώρες μέλη, οπότε να είσαστε σίγουροι ότι θα το λάβουμε υπόψη μας έγκαιρα. Για τις άμεσες ενισχύσεις είναι κατέτος. Και έτσι δεν αναμένουμε καθυστερήσεις. Για την ανάπτυξη φυσικά και πρέπει να έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο έτοιμη, γιατί κάποιες χώρες μέλη θα εξαντλήσουν τα ποσά στο τρέχον πρόγραμμα. Και καλό θα ήταν να μην υπάρχει καθυστέρηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη. Κάποιε χώρε πράγματι δεν θα έχουν πόρου και θα χρειάζονται νέα χρηματοδότηση. Οπότε και αυτό θα το λάβουμε υπόψη μας τις μεταβατικές διευθετήσεις. Ο εισηγητής επίσης ανέφερε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Βεβαίω, η Επιτροπή γνωρίζει ότι το Συμβούλιο το θέλει στο φαρμαστικό, το Κοινοβούλιο το θέλει στα κατεξουσιοδότηση, οπότε εμεί θα φροντίσουμε να περιορίσουμε στο ίμιση ότι είχαμε στην τρέχουσα περίοδο και θα προσπαθήσουμε να είμαστε κάπως στη μέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σίγουρα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις. Έπειτα, ο εισηγητής είπε ότι οι χώρες μέλη θα χρειάζονται νέα συστήματα πληροφορικής. Εδώ πρέπει να πω ότι προσπαθούμε να χτίσουμε στα όσα ήδη υπάρχουν στις χώρες μέλη. Δηλαδή θα συνεχίσουμε με τα σημερινά σώματα διακυβέρνησης, με ό,τι υπάρχει, τους φορείς πληρωμής. Προσπαθούμε δηλαδή να χτίσουμε πάνω σε ό,τι υπάρχει και λειτουργεί. Για τους ελέγχους η πρόταση είναι να έχουν συστήματα ελέγχου οι χώρες μέλη και να χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής γι' αυτό. Χωρίς να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο ελέγχους πρέπει να κάνουν, για παράδειγμα. Γιατί όπως σωστά είπατε, είναι το νέο επίπεδο που βασίζεται στην... σε επιδόσεις. Και οι χώρες μέλη θα πρέπει να το φροντίσουν αυτό, με τη στήριξη βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, και τη 15η Φεβρουαρίου. Γιατί προτείνουμε τη 15η Φεβρουαρίου. Είναι γιατί είναι στον δημοσιονομικό κανονισμό. Το κάνουμε λοιπόν ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να έχει απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει τη δικιά της έκθεση την άνοιξη της χρονιάς. Οπότε μέχρι 15 Φεβρουαρίου χρειάζεται τις εκθέσεις των χωρών μελών. 15 Φεβρουαρίου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις αναφορές των χωρών μελών όχι μόνο για τους λογαριασμούς αλλά και για τις, ε, την επιλογή των δαπανών κατά πόσο είναι επιλέξιμες δηλαδή οι πληρωμές ή όχι. Το ξέρω ότι κάποιες χώρες μέλη λένε ότι αυτό θα είναι δύσκολο. Συγχρόνως όμως το δημοσιονομικό έτος λήγει στις 15 Οκτωβρίου. Οπότε έχουν μέχρι το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο πρέπει να έχουμε τις εκθέσεις τους, να είναι στο σύστημα. Στην κυρία Καρσία Πέρες θέλω να πω για το offsetting ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το offsetting την αντιστάθμιση είναι ένας κανόνας για τους δικαιούχους και για τις χώρες μέλη και για το συντονισμό των πιστοποιητικών φορέων επίσης μπορεί να περιληφθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικές οι διευκρινήσεις και οι εξηγήσεις σας. Κύριε Μπόγκοβιτς, δύο λεπτά ή αν δεν θέλετε. Ένα. Μισό. Ένα λεπτό. Μου φτάνει, μου φτάνει, πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ την Επιτροπή. Η ενημέρωση λοιπόν περιμένει Τα περιμένω τι ε, προτάσει των συναδέλφων, θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία με του σκιώδεις. Μάλιστα λέει η πρόεδρο, ευχαριστώ ακόμα και λιγότερο από ένα λεπτό. Προθεσμία λοιπόν για τι τροπολογίε 12 το μεσημέρι ε, στις 29. Νοεμβρίου, ημέρα 5η, 12 το μεσημέρι, 5η, 29 Νοεμβρίου, προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Γνωμοδότηση. Επί τη προτάσεω κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμων 13.08.2013 και τα λοιπά 13.16 για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Το λόγο έχει ο κύριος Χάουαρτ η Επιτροπή Μεταφορών έχει την ε, έκθεση, σκοπεύει στις 10 Ιανουαρίου να ψηφίσει. Άρα λοιπόν πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας για να προλάβουμε αν θέλουμε βέβαια η γνωμοδότησή μας να επηρεάσει, ε, να κατατεθεί δηλαδή καιρό στην Επιτροπή των Μεταφορών. Άρα σκοπεύουμε η ψηφοφορία για το θέμα αυτό να δεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου έτσι λοιπόν είναι πιο σύντομο ο χρόνος για τι τροπολογίε Έχετε το λόγο κύριε Χάουερθ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια ίσονα προσαρμογή στην νομοθεσία που ελπίζουμε δεν θα χρειαστεί ποτέ να υλοποιηθεί. Δηλαδή, εάν δεν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης, του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουμε ένα τεράστιο κενό στο ε, διάδρομο βόρειας θάλασσης Μεσογείου στο διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Και γιατί, διότι δεν υπάρχει ε, κάποιος τρόπος διασύνδεσης, κάποια λογική διαδρομή για να διασυνδεθεί η υπηρετική Ευρώπη με την νήσο της Ιρλανδίας. Στόχος λοιπόν της πρώτης επιτροπής είναι να οριστεί μια ε, γραμμή ναυσιπλοείας που να ολοκληρώνει έτσι το δίκτυο και ορίζεται το Ρότερνταμ, η Αμβέρσα και η Ζέμπρουχε ως λιμένες α, διασύνδεσης με τους λιμένες του Δουβλίνου και του Κόρκ στην Ιρλανδία. Μπορεί αυτό να φανεί κάπως παράδοξο εκ πρώτης όψεως. Ωστόσο, οι Αύροι και το Ρόσκοφ, λιμένες που μπορεί να θεωρούνται εγκύτεροι, δεν είναι, δεν είναι κατάλληλοι ε, και ούτως ή άλλως ε, οι, οι η Χαβρή ανήκει σε διαφορετικό δίκτυο διευρωπαϊκό από το Ιρλανδικά λιμάνια. Τώρα, είναι μικρό το μέγεθος της αγοράς. Και ίσως και απομακρυσμένη αγορά μπορεί να πει κανείς, επομένως, μπορεί να πει κανείς, επομένως μπορεί να μην επηρεάσει πάρα πολύ μεγάλο όγκο μεταφορών. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι είδους συνέπειες μπορεί να φέρει εάν δεν, ε, το, να μην υπάρξει συμφωνία. Καλέ Ντόβερ Δουνκέρκη θα είναι ήδη ένας από τους ε, δρόμους, από τις διαδρομές που θα έχουν επαρκή προβλήματα, σοβαρά προβλήματα και άρα καλό θα είναι να μην χρειαστεί και το άλλο κομμάτι να αναδιαμορφωθεί και να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ότι ο χώρο του καλέ Ντόβερ και Δουνκέρκης. γιατί δεν υπάρχει καμία, κανένα ιστορικό της διεξαγωγής τελωνιακών ελέγχων στην ε, περιοχή, στη διαδρομή Καλέ ε, Ντόβερ εδώ και τόσο καιρό που κανείς δεν θυμάται πώς θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί ένα τέτοιου είδου, ενός τέτοιου είδους τελωνιακή έλεγχη. Αντίστοιχα λοιπόν θα θέλαμε να αποφύγουμε τα προβλήματα σε περίπτωση χωρίς ε, Brexit στην Ιρλανδία και στη μετάβαση προς τη Βόρειο Ιρλανδία. Επομένως, από την άλλη, αν υπάρξει συμφωνία πάλι θα ε, χρησιμοποιείται ως χερσαία γέφυρα ή νήσος της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Ε, βεβαίως, εδώ έχουμε να κάνουμε με την περίοδο μετά το 2020 και την ολοκλήρωση και της μετάβασης βέβαια που ακόμα δεν έχει διευθετηθεί από το 2021 και μετά που θα καλύπτεται δηλαδή από τον νέο κανονισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει ίσως να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει ίσως να μας ξανααπασχολήσει το πώς θα συνδεθεί η νήσος της Ιρλανδίας με την υπηρετική Ευρώπη και μήπως οι διευθυντήσει για διαδρόμους, για αυτοκινητοδρόμους κτλ. ίσως είναι σκόπιμο να επανεξεταστούν. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank you Σας ευχαριστώ θερμά. Και ευχαριστώ πολύ για το λεπτό εγγλέζικο χιούμορ σας κατά την παρουσίαση της γνωμοδότησης. Εκ μέρους του κυρίου Φαλκάρσελ. Όχι. Δεν βλέπω ούτε άλλους σκιώδη. Α, όχι, να μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμα πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Μια και εμείς έτσι ε, τον Κέρκη και το Καλέ. Παραμένουν λιμένες στο διάδρομο ως λιμένες αναχώρησης. Το καθεστώς αυτό δεν αλλάζει. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο το επισημάνουμε. Καλώ λέει η Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Κόμσμου, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Είναι επακριβέστατη και πλήρης Το θέμα είναι να, λυθούν τα προβλήματα ασυνέχειας τα οποία μπορεί να υπάρξουν στην περίπτωση του ε, Brexit χωρίς συμφωνία επιλέγονται οι τρεις λιμένες οι οποίοι έχουν προς το παρόν ε, αρκετή κυκλοφορία και συνεργασία με την Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ, όλα είναι σαφή, ελπίζω να μπορέσετε να βρείτε μία λύση. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών Είναι 26 Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. 5 το απόγευμα λοιπόν. Έγκριση τώρα των αποφάσεων της, των συντονιστών. Μπορείτε να συμφωνήσετε. Εγώ δεν ήμουν εκεί βέβαια και δεν μπορώ κανονικά να πω πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρακτικά είναι σαφή. Μία παρατήρηση μόνο. Από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μία παρατήρηση. 22 και 21 Ιανουαρίου προβλέπεται να γίνει ψηφοφορία ενώ ο κύριος Σαριμό προτείνει την 3η Δεκεμβρίου. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς ε, Ναι, σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Θα συμπεριλάβουμε λοιπόν την παρατήρησή σας στα πρακτικά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι μπορούμε ε, κάλλιστα να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή χωρίς καθυστερήσεις. Ε, αυτά. Διάφορα, όχι, ωραία. 3 Δεκεμβρίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας από τις 3. Ευχαριστώ πολύ για τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Και κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης για σήμερα.